δήλωση της Επιτροπής και ετήσια έκθεση για τη φορολογία. Ο λόγος στην κυρία Καηλή για τέσσερα λεπτά. Και να χαιρετήσω και τον Αντιπρόεδρο Μοσκοβισή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Καηλή. Uh, Συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, από τις βασικότερες προκλήσεις της ε, ετήσιας έκτης για τη φορολογία ήταν ε, να εκθέσει μια πιο πολιτική άποψη για το θέμα και όχι απλώς να ακολουθήσει την πεπατημένη του τίποτα δεν έχει αλλάξει. Και μάλιστα ε, η εμφάνιση της υπόθεσης Λίξκ κατά την εκπόνηση ανέδειξε την ανάγκη μιας υπεύθυνης πολιτικής ανάπτυξης. Έπρεπε να λάβουμε πολιτική θέση και όχι να προσπίθουμε ότι τίποτα δεν συνέβη. Και μάλιστα η ετήσια εκθεσία αποτελεί το βασικό εργαλείο της ΕΚΟΝ για τα φορολογικά θέματα. Και μάλιστα το ενδιαφέρον, το ζωηρό ενδιαφέρον φάνηκε από την πληθώρα των τροπολογιών που ζητούν συγκεκριμένο χειρό πολιτικό μήνυμα. Πολλές προτάσεις υποβλήθηκαν, για παράδειγμα θέματα ε, να αποκατασταθεί κοινωνική δικαιοσύνη στις φορολογικές πολιτικές, ε, να φορολογηθεί το κεφάλαιο, ε, το, οι τα μερίσματα, επίσης να ελεγχθούν κάποια χρηματοοικονομικά μέσα που διευκολύνουν τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή. Επίσης, το θέμα της, ε, του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι πολύ δημοφιλές. Πολλοί ε, συνάδελφοι ζήτησαν να, ενισχυθεί και να χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες αυτές για να ε, ενισχυθεί το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ταμείο για τις Κλιματικές Αλλαγές, είτε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Επιπλέον, από τη συζήτηση φάνηκε η μόνιμη ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το φόρο εταιριών, ιδιαίτερα την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις και τις ελάχιστες ε, φορολογικές συνεισφορές των εταιριών. Πολλές προτάσεις συνέδεσαν τη φορολογία με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ε, κατέθηκαν τροπολογίες για τη φορολογική μεταχείριση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βέβαια, ακόμη έχουμε διαφωνία μεταξύ αυτών που είναι υπέρ του συντονισμού και εκείνων που είναι υπέρ της εναρμόνισης. Βέβαια, ο συντονισμός ε, δεν έχει επιτύχει, φάνηκε από το Leaks και το LuxLeaks. Επίσης, ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την εναρμόνιση σε φορολογικά θέματα, χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και άλλους τρόπους ε, για να μπορέσουμε να επιβραβεύσουμε τους έντιμους φορολογούμενους. Επίσης, προσπαθήσαμε με την αναζήτηση συμβαστικών λύσεων να υιοθετήσουμε υπεύθυνη θέση, να καταπολεμήσουμε τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, το φορολογικό, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και να μειώσουμε το φορολογικό χάσμα. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα για τις φορολογικές πολιτικές που θα ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και θα στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης θα πρέπει να αντιληφθούμε τις κοινωνικέ συνέπειε των φορολογικών πολιτικών, ιδιαίτερα για τους οικονομικά πιο ευάλωτους συμπολίτε μας. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε και αργότερα ε, σε κοινέ πρωτοβουλίε οικονομικής πολιτικής. Για παράδειγμα, θα πρέπει να έχουμε κοινό ορισμό των φορολογικών παραδείσων, ε, επίσης κυρώσεις για τους ε, δράστες φορολογικών απατών, να αποφύγουμε ε, την μεταφορά των κερδών για πιο ευνοϊκή φορολόγηση και το, το θέμα των, φορο, των συναλλαγών, του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επίσης το θέμα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και της ε, αποφυγής ε, αδιαφανών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρονται γι' αυτό και Ευρωπαίοι πολίτες ε, να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ξεκάθαρη θέση κατά οποιοδήποτε αδιαφανούς πρακτικής που ενισχύει την ασάφεια και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό. Επίσης, θα, με τη διαφάνεια θα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και την φοροδιαφυγή. Πια δεν μπορούν οι τράπεζες να αρνούνται δημοσίευση ε, ε, κάποιων στοιχείων με πρόσχημα το βιομηχανικό ή εμπορικό απόρριτο. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε σαφή μέτρα ε, και συνέπειες συγκεκριμένες για τους ε, παραβάτες όλων αυτών των διατάξεων. Η ετήσια φορολογική έκθεση ε, έχει μία συνεπή θέση και αποτελεί τη βάση για μία φορολογική πολιτική που θα είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις, προς το περιβάλλον και τους φορολογωμένους. Ευχαριστούμε κυρία Καηλή. Λυπάμαι, σα άφησα λίγο χρόνο παραπάνω μεν, αλλά θα πρέπει να είμαι πολύ αυστηρή με του υπόλοιπου. Πρέπει να έχουμε πολύ λίγο χρόνο για τι τόσε συζητήσει μα, γι' αυτό δίνω το λόγο στον κύριο Μοσκοβισή. Ε, κύριε Μοσκοβισή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι και κυρίες, ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να συζητήσουμε την φορολογία στην Ευρώπη. Η έκθεση που συζητάμε σήμερα κάνει μια διάγνωση την οποία συμμερίζομαι πλήρως. Το πανόραμα της φορολογία των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων είναι και μη αποτελεσματικό και μη διαφανές. Οι κανόνες των κρατών μελών θέτουν θεμελιώδη προβλήματα για όλη την Ένωση. Πρώτον, οι φορολογικοί κανόνες πολύ συχνά κατακαιρματίζουν την ενιαία αγορά ούτως ώστε οι περισσότερες ευρωπαϊκές ή ξένες επιχειρήσεις δεν έχουν πλήρη ε, πρόσβαση και πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια που του δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του. Και οι φορολογικέ αρχέ δεν έχουν τη δυνατότητα, όλο και λιγότερο έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν το φόρο που θα έπρεπε. Ορισμένοι φορολογούμενοι κάνουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό για να υποφεληθούν από τι ασυνέπειες και τι διαφορέ των φορολογικών συστημάτων και επιπλέον πρέπει να σημειώσουμε ότι τα κράτη-μέλη, ακόμη και αυτά, κάνουν υπερβολικό ανταγωνισμό για να προσελκύσουν τις πιο ε, ευκίνητες βάσεις φορολόγησης. Το σύστημα λοιπόν αυτό είναι άδικο και βοηθάει τους πιο ισχυρούς σε βάρος όλων των υπολείπων. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε κάτι τέτοιο γιατί είναι απαράδεκτο. Και η ίδια η αποδοχή της φορολογίας μειώνεται και αυτό είναι το βασικό στοιχείο του κοινωνικού συμβολέου μεταξύ των αρχών και των πολιτών. Είναι λοιπόν κρίσιμη η κατάσταση. Και χρειαζόμαστε, χρειαζόμασταν επίγουσα και ευρία δράση. Οι στόχοι μου είναι οι ίδιοι με τους δικούς σας. Πρώτα απ' όλα Πρέπει να επανέλθει η φορολογική δικαιοσύνη και στην Ένωση και στα κράτη-μέλη, να δημιουργήσουμε επιτέλου πραγματική, μια πραγματική εσωτερική αγορά για φορολογικά θέματα που να είναι διαφανή και προβλέψιμη για να μπορούν να επενδύσουν οι εταιρείε και να επανέλθει η εμπιστοσύνη για του καταναλωτές. Και η φορολογία μα πρέπει να είναι στο, στην υπηρεσία τη πολιτική μα, Είτε είναι για την φορολογική ατζέντα ή για την Ένωση ενέργεια. Υπάρχουν λύσει. Ορισμένε τι ξέρουμε ήδη εδώ και χρόνια. Αλλά για να τι εφαρμόσουμε θα χρειαστεί αποφασιστικότητα από πλευρά όλων. Πρώτα απ' όλα από τα περισσότερα κράτη-μέλη που θα έχουν τελευταία λέξη γι' αυτό. Και θα πρέπει να συμφωνήσουν για τι φιλόδοξε λύσει που προτείνουμε. Ο πρόεδρο τη Επιτροπής έθεσε την καταπολέμηση τη φοροαπάτης και της φοροαπαλλαγή ως απόλυτη προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα επιμείνω σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω ξέρετε, μόλι πήρε μια σειρά από ισχυρών μέτρων για να βελτιωθεί η φορολογική διαφάνεια στην Ένωση Πρώτα απ' όλα είχαμε την πρόταση οδηγίες για την ανταλλαγή πληροφοριών, για τις φορολογικές συμφωνίες, ούτως ώστε να έχουν όλα τα κράτη-μέλη πληροφορίες για τις επιπτώσεις των αποφάσεων των εταίρων τους στη δική τους βάση φορολόγησης. Και επίσης δεσμευόμεθα ιδιαίτερα να προωθήσουμε την ε, διαφάνεια και πέρα αυτών των φορολογικών συμφωνιών, το ruling, για να είμαστε πρωτοπόροι σε παγκόσμια κλίμακα για το τομέα αυτό, όπως προτείνεται, θα μπορούσαμε μέσω αυτής της, ε, όπως λέτε στην έκθεση, να επεκτείνουμε τις υποχρεώσεις για μερικές μεγάλες επιχειρήσεις να γνωστοποιούν ε, ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού τους αναχώρα. Αυτό να το δούμε ως Επιτροπή με το Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη διαδικασία, θα πρέπει να κάνουμε πιο σε βάθος ανάλυση, αλλά θα εργαστούμε ταχύτατα για να γίνει αυτή η ανάλυση, γιατί είναι προϋπόθεση για να πάρουμε κοινέ θέσει κατόπιν. Το θέμα του τόπου όπου πρέπει να φορολογούνται τα κέρδη είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει από τη μία μεριά η Ευρωζώνη και από την άλλη η ενιαία αγορά με 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Έχουμε τους κανόνες μας, τις προτεραιότητές μας, τους στόχους μας. Η Ένωση μπορεί να βασιστεί και στην πολύ καλή εργασία του ΟΟΣΑ, αλλά όχι μόνο σε αυτήν. Γι' αυτό το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2015 λέει ότι υπό το φως των παγκοσμίων εξελίξεων θα υποβάλει πρόγραμμα δράσης για την φορολογία των εταιριών στην ενιαία αγορά. Τα κέρδη θα πρέπει συστηματικά να φορολογούνται εκεί που προκύπτουν. Έτσι θα, ξεκινήσει, επανέλθει η συζήτηση για το πρόγραμμα άξης, ούτω ώστε να αρμονίσουμε την βάση φορολογηση για διάφορε διαμεθοριακές επιχειρήσει στην Ένωση. Αυτό θα βοηθήσει να γίνει πιο ανταγωνιστική η αγορά, αλλά παράλληλα θα περιορίσει τι δυνατότητε οι διάφορε εταιρείε να κάνουν διάφορε λαθροχειρίε Και θα υπάρξουν και, και, προ, και πιο βράχη πρόθεσμα μέτρα για να εφαρμόσουμε ως Ένωση τις παγκόσμιες αποφάσεις, για παράδειγμα, σε επίπεδο G20 και η Επιτροπή θα εγκρίνει λοιπόν το πρόγραμμα δράσης πριν το καλοκαίρι, αρχές Ιουνίου. Είμαι πεπισμένος ότι το σώμα σας μέσω των Επιτροπών για τη Φορολογία και την ΕΚΟΝ θα συμβάλλει στην προετοιμασία αυτού του προγράμματος δράσης. Να πω δύο λόγια τώρα για δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θέλουμε να υπάρξει ένα φιλόδοξο σχέδιο σε εθνικό επίπεδο είναι κάτι που συμφωνούμε με εσά, όπως το είπε και ο πρόεδρος Γιούγκερ. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τις φορολογικές ε, μεταρρυθμίσεις για να φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι υποφελήθηκαν από τις τελευταίες εξελίξεις και να μειωθεί ε, ο φορολογικός φόρτος της εργασίας. Και τονίζω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν εθνικό φόρο επί των χρηματοστοιχών συναλλαγών στη Γαλλία από το 2016. Και οι χώρε μέλη τη ενισχυμένη εργασία είπαν ότι οι εθνικοί τέτοιοι φόροι πρέπει να βασίζονται στην πιο ευρεία βάση φορολόγηση με χαμηλά βεβαίω επιτόκια. Λαμβάνοντα υπόψη την επίπτωση στις, ε, στην πραγματική οικονομία. Οι υπηρεσίε τη Κομισιόν θα συνεχίσουν να προσφέρουν τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη για να καταλήξουν σύντομα σε μια συμφωνία με βάση την πρόταση επιτροπή και με πνεύμα συνεργασία. και θετικό. Για του έμεσους φόρους τώρα. Υπογραμμίζω ότι η Κομισιόν κατά τη θητεία τη θα υποβάλει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις, για να βελτιωθεί η λειτουργία του ΦΠΑ, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να καταλήξουμε σε ένα οριστικό καθεστώς του ΦΠΑ. Η Κομισιόν είναι υπέρ μιας ε, συνολικής άποψης και όχι διάφορα μέτρα ad hoc ε, κατακαιρματισμένα γιατί κάτι τέτοιο κατά τι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυνεπεί λύσει. Ξέρουμε πώ γίνονται αυτά. Ή μπορεί να μην καταλήξουμε σε καμία λύση. Και αυτό βεβαίω ε, θα αφορά και του συντελεστέ του ΦΠΑ. Ευχαριστώ την κυρία Καλή για τη θαυμάσια εργασία τη. Είμαι στην διάθεση του Κοινοβουλίου για να προχωρήσουμε μαζί σε αυτά τα τόσο ουσιώδη θέματα. Και θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με την Ειδική Επιτροπή για τι ε, φορολογικέ αποφάσει σε πνεύμα συνεργασίας και διαφάνειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, για την συμβολή σας και τώρα αρχίζουμε τον κατάλογο των αγορητών για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Τόλογιαν. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να καλωσορίσω την νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το τα μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια δηλαδή. Είμαι βέβαιος ότι με την εισαγωγή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις, ε, φορολογικέ συμφωνίε, θα... και τις φορολογικές αποφάσεις θα ε, ενημερώνονται ευθύ αμέσω οι πολίτε μα, διότι τα κέρδη από ε, την φορολογία θα πρέπει να συγκεντρώνονται εκεί όπου έχουν πραγματοποιηθεί τα κέρδη. Δεν μπορεί να κλειτώνουν τη φορολόγηση κάποιοι λόγω της δημιουργικής λογιστικής. Εδώ λοιπόν καλωσορίζω όσα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη φοροδιαφυγή και την ε, φοροαποφυγή και να ευχαριστήσω και την κυρία Καϊλή για την έκθεσή της όπως και άλλοι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκα πολύ αποτελεσματικά για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση για μια πολύ σημαντική ιδέα εδώ. Συνεργαζόμαστε στενά σε επίπεδο κρατών μελών και μέτρητα κράτη. Εφόσον ενταθεί αυτή η συνεργασία θα επιτύχουμε πραγματική πρόοδο για την καταπολέμηση της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής και θα την διαφυγή των κερδών στις χώρες και, όχι στις χώρες από αυτές όπου έχουν πραγματοποιηθεί. Ναι, ξέρετε, αλλά έχουμε μια μισή ώρα καθυστέρηση, συνάδελφοι, οπότε θα κάνω την εξή πρόταση. Δεν θα έχουμε γαλάζιες κάρτες, διότι πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν να παρέμβουν με γαλάζια κάρτα, αλλά ελπίζω να καταλάβετε εδώ την ε, απόφασή μου. Ε, περνάμε αμέσως στην επόμενη μελήτρια για δύο λεπτά, η κυρία Φερέιρα. Κύριε Επίτροπε, η χώρα μου, η Πορτογαλία, όπως ε, και πολλές άλλες ξέρει, ότι υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν από την κρίση. Ε, πρέπει με δυσκολία να βρουν κάποιο δάνειο και να πληρώσουν 23% φόρο για τη κέρδη τους. Ενώ μεγάλες πολυεθνικές, όπως Amazon, Starbucks, ε, καταφέρνουν ε, ανεξέλεγκτα να πληρώνουν φόρους που ξεπερνούν μόλις το 1% παίζοντας μεταξύ των ε, φορολογικών ανισοτήτων των κρατών μελών. Η χώρα μου δεν επέτυχε αρκετά φορολογικά έσοδα για να καλύψει τα ελλείμματα στην εκπαίδευση, την υγεία ή για να αντιμετωπίσει την κρίση και με κίνδυνο να επιβληθεί πρόστιμα, ε, πρόστιμα 5% του ΑΕΠ για την ε, πλημελή συμμορφωσή μας με τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης. Ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Πορτογαλίας που θα μπορούσαν με την φορολογική του συμβολή να οδηγήσουν στην εξισορρόπηση των δημοσιονομικών τελικά, ε, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, ε, μπορούν να μετακινήσουν τη φορολογική τους έδρα σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο για να υποφεληθούν από όσα ισχύουν. Ε, για εταιρείε που λειτουργούν στην ίδια αγορά και σε, ένα, σε μια ζώνη ενιαίων νομίσματος δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για, για τις ίδιες εταιρείε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, επιμείνει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφόρων μεταξύ των κρατών μελών και θα συγχαρώ για αυτό τον κύριο Επίτροπο. Όμω δεν αρκεί. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για να καταπολεμήσουμε και του φορολογικού παραδείσου και την δυνατότητα των ε, ε, μεγάλων εταιριών να εκμεταλλεύονται τι φορολογικέ διαφορέ μεταξύ χωρών και να απαιτήσουμε να υπάρξει πρόοδος, επιτάχυνση στην εξέταση των θεμάτων αυτών. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι πλήρως αποφασισμένο να συμμετάσχει σε αυτή τη νέα ε, νοοτροπία στην φορολογική μεταχείριση και ελπίζουμε πέραν της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, πέραν της στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχουμε το ίδιο πνεύμα σύγκλησης και συνεργασίας και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι πολίτες το απαιτούν και αυτήν την απόκριση οφείλουμε να τους δώσουμε. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Κούσμιουκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχουμε ε, κάποιες, κάποια στοιχεία εναρμόνισης, όπως το ΦΠΑ, μη εναρμόνισης, όπως φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ε, και εξαιτίας αυτής της αναντιστοιχίας υπάρχουν πολλά αρνητικά φαινόμενα δύο την Ε, η, ήδη έχουμε εκατομμύρια, ε, ε, εκατομμύρια ευρώ που χάνονται από τα εισοδήματα του ΦΠΑ εξαιτίας της μη εναρμόνισης. Επίσης έχουμε ε, φορολογικές απάτες τύπου καρουζέλ ε, μεταξύ επιχειρήσεων διαφόρων χωρών, χωρίς, με εικονικές όμως συναλλαγές και έτσι διαφυγή, φοροδιαφυγή σε ό,τι αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Επίσης, ε, μερικές φορές ε, και η επιστροφή του ΦΠΑ δεν γίνεται με σωστό τρόπο. Έχουμε μεγάλη απώλεια φορολογικών εσόδων. Επίσης, ε, μεγάλοι όμιλοι και πολυεθνικές χρησιμοποίησαν φορολογικό ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, 4 δισεκατομμύρια έχασε η Πολωνία από τέτοιους φορολογικούς, φορολογικές μυστικές συμφωνίες που ε, Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σας διακόψω. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή για τις συζητήσεις αυτές. Θα, είμαι πολύ αυστηρή, πρέπει να παραμένετε στα του χρόνου σας. Δεν μπορώ καθόλου να κάνω εξαιρέσεις. Θα δώσω το λόγο στην ε, επόμενη μιλήτρια, την κυρία Βανίβαν Χόιζεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, πριν από μερικά χρόνια είχα δηλώσει ότι με ενδιαφέρουν τα φορολογικά θέματα και τότε με κοιτούσαν με ήκτο μερικές φορές γιατί το θέμα αυτό το έκρινα πολύ ε, βαρετό, κουραστικό. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει και από πολιτική άποψη για πολλούς και διάφορους λόγους. Ε, με τη LuxLeaks ε, τα φορολογικά θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής, ακόμη και του απλού πολίτη. Ε, μερικές φορές οι απλοί πολίτες έχουν την αίσθηση ότι καταβάλουν πολύ περισσότερους φόρους από, από τις μεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως πολυεθνικές που καταφέρουν με διάφορες φορολογικές συμφωνίες να απαλλαγούν από την καταβολή των φόρων. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποια βήματα, αλλά να ξέρουμε γιατί μιλάμε και να χρησιμοποιούμε τους ίδιους όρους, τους ίδιους ορισμούς και την ίδια ορολογία. Γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή, ε, την φοροαποφυγή. Τι θα πει φορολογικό παράδεισος, γιατί δεν έχουμε ένα κοινό ορισμό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε για να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για ενίσχυση της διαφάνειας. Επικροτούμε την αξιέπαινη αυτή προσπάθεια, γιατί για να ξέρουμε γιατί μιλάμε χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα διαφάνεια. Και έχω και μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε όλοι ότι το πρόβλημα έχει παγκόσμιες διαστάσει. δεν περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Οπότε κύριε Επίτροπε, πώς θα διαπραγματευτεί το θέμα της διαφάνειας με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Ευχαριστώ και πιστεύω ότι τήρησα το χρόνο μου κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό τώρα η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ο τομέας της φορολογικής πολιτικής ε, είναι ένας τομέας όπου υπάρχουν πολλές αδικίες και ανισότητες. Είδαμε τα τελευταία χρόνια με την κρίση να υπάρχουν αυτά τα φοβερά μέτρα λιτότητας που έπληξαν την ανταγωνιστικότητα προκειμένου να συγκεντρωθεί περισσότερο κεφάλαιο στα ίδια χέρια και ως προς το κέρδος και ως προς το ωφέλη. Και με την δημοσιονομική πίεση φτάσαμε στο απίστευτο ε, σημείο αυτό υποβάθμισης και της απασχόλησης και της κατανάλωσης Έχουμε λοιπόν καταστρεπτικές συνέπειες, κυρίως για την περιφέρεια της Ευρωζώνης. Η συνέπεια είναι ότι η κατανομή του πλούτου και του κέρδους είναι πλέον περισσότερο άδικη από ό,τι Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε και τα σκάνδαλα που προέκυψαν με την φοροαπάτη και τη φοροδιαφυγή και βλέπουμε ότι το LuxLeaks είναι απλώς η αιχμή του δόρατος εδώ πέρα, ε, η κορυφή μάλλον του παγόβουνου θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι χάνεται ένα 3 ευρώ λόγω των ε, ε, ατασταλιών και των παράνομων φορολογικών πρακτικών στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να μην ε, επίσης να δούμε ότι μετακίνησαν τι έδρε του προ την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο 20 μεγαλύτερε πορτογαλικέ εταιρείε για να γλιτώσουν ακριβώς τη φορολόγηση. Εδώ η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση με μέτρα που ήδη υπήρχαν από το 77 ε, δεν τα υλοποίησε και τώρα μιλά για διαφάνεια και φορολογική ενοποίηση. Μου φαίνεται ε, ε, κάτι παράλογο αυτό, διότι διαφάνεια είναι ένα δημόσιο αναφέρεται δικαίωμα. Ευχαριστούμε και τώρα για τρία λεπτά η κυρία Σκοτ Κάτω. Για πολλούς τον τελευταίο χρόνο ο φόρος έχει γίνει θέμα μεγάλο ενδιαφέροντος. Επειδή οι επιχειρήσεις και οι πλούσιοι έχουν βρει όλο και πιο περίπλοκους τρόπους να μην πληρώνουν ό,τι θα έπρεπε, έχει γίνει ενδιαφέρον το θέμα. Και οι κυβερνήσεις δεν έχουν το αναγκαίο εισόδημα και δεν μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις για υποδομές, για τους ευάλωτους. Φτάσαμε σε ένα σημείο που είναι ζωτικό για την προστασία της πολιτισμένης κοινωνίας μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Η φοροδιαφυγή υπονομεύει και την ενιαία αγορά οι διαμεθοριακές εταιρείε κάνουν κυβερνήσεις, ε, κάνουν συμφωνίες ε, προτιμησιακές με τις κυβερνήσεις που δεν θα μπορούσαν να τις κάνει καμία μικρομεσαία που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Οι πράσινοι που είναι υπέρ της τοπικής οικονομίας θέλουν η ολοκλήρωση της ενέργειας αγοράς να γίνει με δίκαιη φορολογία παντού στην Ένωση για να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ μικρομεσαίων και πολυεθνικών. Τον περασμένο Νοέμβρη όταν έγινε γνωστό τις σκανδαλώδη συμφωνίες είχε κλείσει ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ ως πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ζητήσαμε, έγινε μία πρόταση για να γίνει μορφή σε ολόκληρη την Επιτροπή. Αλλά παρά τις αμφιβολίες που είχαμε για κάποιους επιτρόπους, εμείς θεωρούμε και θεωρήσαμε τότε ότι πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία. Να την αξιοποιήσουν λοιπόν, αλλιώ να φύγουν. Είδαμε τώρα τι προτάσει τη Κομισιόν. Δεν θα σα εκπλήξει ότι μα απογοήτευσαν ιδιαίτερα. Η πρόταση για την ανταλλαγή προφορών μεταξύ κρατών μελών είναι αναγκαία. Την καλωσορίζουμε. Αυτό διευκρινίζει μια υποχρέωση που ισχύει υποτίθεται από το 70 αλλά ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί. Αν είχε εφαρμοστεί θα έχει διασφαλίσει ότι αυτέ οι σκανδαλώδει φορολογικέ συμφωνίε δεν θα μπορούσαν να μείνουν κρυφέ. Όμω είναι μόνο ένα μέτρο. Πολλά άλλα πρέπει να εισαχθούν για να βελτιωθεί η διαφάνεια. Χαίρομαι λοιπόν για τις κατηγορηματικές δηλώσεις που έχουν γίνει για το θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού και της φόρου αποφυγής που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση. Ιδιαίτερα η επανειλημμένη έκκληση για κοινό και υποχρεωτικό σύστημα φορολογικής βάσης για τις εταιρείε. Και καλωσορίζω και την Ειδική Επιτροπή που κάναμε για να, για να διερευνήσει αυτά τα θέματα. Αλλά ως πράσινη, γιατί φέτος που θα γίνει η συνάντηση στο Παρίσι, οι προτάσει που κάναμε για να σταματήσουν οι εξαιρέσει για, την αεροπορική, για τον αεροπορικό κλάδο και οι άλλες επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα απορρίφθηκαν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αν αξιοποιήσουμε στρατηγικά τη φορολογία μπορούμε να δώσουμε κίνητρα ούτω ώστε οι κοινότητέ μα να έχουν ένα μέλλον όπω θα το θέλαμε για τα παιδιά μα. Βιώσιμο και δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσάνι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Υπόθηκε ότι μετά το σκάνδαλο Κλικς κάτι θα έπρεπε να γίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχολείται πολύ σοβαρά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ε, φόροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Ε, που υπάρχει σε που ανταπαντάται σε πολλά κατημέλη. Όλοι όμως ξέραμε τι θα γίνει. Ο κύριος Γιούνκερ με τόση εμπειρία τόσα χρόνια στο Λουξεμβούργο είχε εγγυηθεί ότι σε πρώτο πρόσωπο θα αναλάβει ο ίδιος την δράση κατά των φαινομένων αυτών. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε λοιπόν ότι απλώς ε, πρόκειται για μια θεατρική παράσταση επιτρέποντας ε, στα κάτι μέλη να συνεχίσουν τις ίδιες πρακτικές με ό,τι μέσα χρησιμοποιούσαν ω τώρα. Και το ίδιο και με τι προτάσει του Επιτρόπου Μοσκοβισή την περασμένη εβδομάδα. Ε, ουσιαστικά την κακή πίστη και την ανικανότητα δεν την αντιμετωπίζουμε. Τα συστήματα αυτά, είτε είναι διαφανή είτε όχι, ουσιαστικά είναι νομότυπα. Επιτρέπουν να λαμβάνονται μεμονωμένε αποφάσει και τελικά μια απλή υποχρέωση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών δεν εξασφαλίζουν τίποτα. Δεν έχουν πρόσβαση πολίτε τα ε, έγγραφα αυτά. Δεν είναι αυτό λοιπόν αυτό που χρειαζόμαστε. Το θέμα είναι ένα ένα και μόνο. Πρέπει να αλλάξουν οι κανόνε, διότι αν, αυτοί, αν αυτέ οι διαδικασίε συνεχίσουν να είναι νομότυπε, η κατάσταση δεν θα αλλάξει ποτέ. Όλο ένα θα συζητάμε για περισσότερη και μεγαλύτερη διαφωνία με συνεργασία, χωρί να επιλύεται κανένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, ζητώ εγώ και άλλοι 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε, εάν επιτέλου υπάρχει πολιτική βούληση για να, για να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα. Τι νόημα έχει να μιλάμε για αλληλεγγύη στην Ευρώπη, να επιτρέπονται αυτέ οι πρακτικέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριο Κόρβιν Μίκε. Ευχαριστώ. Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαφορετικότητα, η πολυμορφία. Για κάθε θέμα απαιτείται δηλαδή απολυταρχική εναρμόνιση αν κάποιος από την Πορτογαλία λέει ότι οι άνθρωποι φεύγουν προς την Ολλανδία, ε, ας μειώσουν το φορολογικό τους, το φορολογικό τους συντελεστή, ώστε να έχουμε αντίθετη μετακίνηση από την Ολλανδία προς την Πορτογαλία. Θα πρέπει να δώσουμε ανάψματα στις κυβερνήσεις για ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων, μεταξύ των ε, ε, πολιτών. Αλλά βλέπουμε ότι στην αίθουσα επικρατεί η απολυταρχική άποψη ότι όλα πρέπει να είναι ενιαία και ομοιόμορφα εναρμονισμένα. Θα πρέπει να καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Sorry, colleagues. Please, we'll παρακαλώ. Ενάμιση λεπτό. Ο κύριος Μπάλτς. Καλωσορίζουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τα πρώτα βήματα για την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Καιρός ήταν αλλά δεν επαρκούν. Σωστό και απόλυτα αναγκαίο κατά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών να επιμείνουμε. Πρέπει να είναι υποχρεωτικό και τακτικός αυτό ο έλεγχος και επαληθεύσιμο. Είναι σωστό και απόλυτα αναγκαίο. Οι παγκόσμιες ε, συμφωνίες του ΟΣΑ για την φορολογική διαφάνεια να εφαρμοστούν. Και πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις γι' αυτό. Και πρέπει οπωσδήποτε η Κομισιόν να, ε, να δημιουργήσει αυτή την κοινή βάση φορολόγηση των επιχειρήσεων. Και επίσης, σωστό και αναγκαίο, είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της ομάδας για τον κώδικα διοντολογίας και να ελέγχουμε τις πληροφορίες που μας δίνουν οι πολυεθνικές. Αλλά δεν είναι αναγκαίο να κάνουμε μια νέα γραφειοκρατία. Να θέσουμε δηλαδή μεγάλο ε, γραφειοκρατικό άχθος πάνω στις επιχειρήσεις. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια επίθεση επενδύσεων, καινοτομίας και απασχόλησης. Εάν επιβάλλουμε λοιπόν σε όλες τις επιχειρήσεις τρομερές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, αυτό θα έχει τρομερό κόστος, πρέπει να είμαστε αναλογικοί γιατί αλλιώς θα καταστρέψουμε την όλη προσπάθεια. Οπότε η υποχρεωτική επιβολή υποχρεώσεων δεν μας βρίσκει συμφώνους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Δύο λεπτά ο κύριος Ζήμων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αθέμητες αλλά όχι παράνομες πρακτικές υπάρχουν ε, στην Ένωση και τις έχουμε ανεχθεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι πολίτες δεν το γνώριζαν αυτό. Και τώρα μόνο πριν από μερικούς μήνες όταν προέκυψαν τα θέματα του LuxLeaks καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Οι πολίτες διερωτώνται πώς είναι δυνατόν οι μεγάλες πολυεθνικές σε βάρος ε, τρίτων να διαπραγματεύονται το φορολογικό συντελεστή τους. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό, αν θέλουμε αυτές οι αθέμητες πρακτικές να ε, συνεχιστούν, χρειαζόμαστε διαφάνεια. Και γι' αυτό η πρωτοβουλία που ξεκίνησε τώρα η Κομισιόν είναι ένα πρώτο λιθαράκι. Δεν θα είναι δυνατόν να αποφεύγουν τι υποχρεώσει του εάν είναι υποχρεωμένη η ανταλλαγή προφοριών μεταξύ κρατών μελών. Ωστόσο, υποχρεώσει είχαμε επιβάλει και στο παρελθόν. Πρέπει να προσέξουμε ότι στο μέλλον οποιοδήποτε δεν τηρεί αυτές τις υποχρεώσει θα τιμωρείται. Μόνο όποιο φοβάται τι συνέπειε θα συμμορφωθεί. Πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν από αυτό. Είναι καλό που η Κομισιόν τώρα προτείνει να υπάρχει ένα κεντρικό μητρό όπου να αναφέρονται όλες αυτές οι φορολογικές συμφωνίες. Όμως αυτό που είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι συμφωνίες των επιχειρήσεων να περιέχονται σε αυτό το μητρό και αυτό το μητρό να μην ε, ανοιχτό μόνο για τα κράτη-μέλη αλλά με βεβαίω ε, ε, και στην κοινή γνώμη με τις αναγκαίες ε, προστασίες προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να είναι δημόσιο αυτό το Μητρό. Καλωσορίζουμε το, το Κομισιόν σκοπεύει να υποβάλει το δεύτερο πακέτο φορολογικής διαφάνειας για μια κοινή βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Όμως, θέλω να τους ενθαρρύνω να δουν τι μπορούν να κάνουν και περαιτέρω. Δηλαδή να δούμε το θέμα μέσω μια έκθεση χώρα ανά χώρα για να δούμε πού πληρώνουν οι πολυεθνικέ του φόρου του. Η διαφάνεια είναι το πρώτο βήμα ούτω ώστε το αθέμητο να γίνει και παράνομο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η φοροδιαφύγη χρησιμοποιώντας και νόμιμες μεθόδους αλλά και παράνομες μεθόδους κοστίζει πάρα πολύ εις βάρος των προϋπολογισμών μας. Γι' αυτό με ικανοποίηση βλέπω την πρωτοβουλία της Επιτροπής με μια πρόταση που είναι το πρώτο βήμα για να μπει τάξη επιτέλους σε αυτόν τον τομέα με την υποχρεωτική ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Καηλή, συγγήτρια, διότι υπέβαλε, η κυρία Καηλή που υπέβαλε μια πολύ ισορροπή έκθεση. Είναι ένα θέμα επίμαχο και θα ήθελα να τοποθετηθώ. Στο εδάφιο 25 η κυρία Καηλή προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει μία βάση για την φορολογία, ελάχιστη φορολογική βάση, για να πετύχουμε να περιορίσουμε τον μη νόμιμο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Θεωρώ ότι είναι κακή ιδέα για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, τα κράτη-μέλη έχουν ένα συγκεκριμένο ξεχωριστό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Κάποια κράτη μπορούν να προσφέρουν καλές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εταιριών τους, άλλα κράτη δεν έχουν τόμως υποδομέ υποδομές και τα μέσα Γι' αυτό δεν θα ήταν πολύ επαρκές να ε, καθορίσουμε μια ελάχιστη φορολογική βάση. Ίσως υπάρχουν και κράτη-μέλη που δεν μπορούν να είναι σε θέση να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες ε, στις επιχειρήσεις τους. Δεύτερον, πρόκειται και για ένα πολιτικό πρόβλημα. Άσχετα ποια θα είναι τα πολιτικά κόμματα για το, ε, τον καθορισμό της φορολογικής βάσης, δεν πρέπει να καταλήξουμε σε μια τέτοια εκλογική αντιπαράθεση. Ευχαριστώ. Και τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, Θυμάμαι που ήμουν εδώ πριν από πέντε μήνες αμέσως μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου των Leaks Και πριν από δύο μήνες συζητούσαμε άλλο σκάνδαλο, τα Swiss Leaks. Ποια ήταν λοιπόν η πρώτη ανταπόκριση της Κομισιόν. Χαιρετίζω τα μέτρα που συμμενέστησε για τις φορολογικές διευθετήσεις, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερη δράση αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις ευχές των πολιτών μας. Με ανησύχησε γιατί το ότι ήταν τόσο ψυχρή η ανακοίνωση της ε, Κομισιόν. Ελπίζω να μας αφήσει να συνεχίσουμε τη δική μας εργασία για την προώθηση αυστηρότερων μέτρων και το κοινό, οι πολίτες θέλουν άμεση δράση. Ήδη έχουμε στοιχεία ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από τις εκθέσεις αναχώρα. Ξέρουμε μάλιστα ότι θα έχει θετικές επί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αυτή τη στιγμή δεν ανταγωνίζονται η μια την άλλη ισότιμα. Ελπίζω λοιπόν η Κομισιόν να υποστηρίξει το αίτημά μας για εκθέσεις αναχώρα επιγόντως. Επίσης υπάρχουν και άλλα αιτήματά μας. Όχι μόνο το CCCTB, αλλά και την γενικότερη πάταξη της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής με καλύτερο ορισμό και των φορολογικών παραδείσων. Ευχαριστώ για ένα λεπτό τώρα. Ο κύριος Βαντερκίντελάρα. Πρόεδρε, συνάδελφοι, όλοι θέλουμε μια πιο υγιή ατμόσφαιρα, αλλά για να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός πρέπει οι κανόνες να είναι ισότιμοι για όλους και διαφανείς. Η δέσμη φορολογικής διαφάνειας που προτείνει η Κομισιόν είναι ένα σημαντικό βήμα και μας επιτρέπει να δούμε τι συμβαίνει και με τη φοροαποφυγή αλλά πρέπει να έχουμε πραγματικά όπλα για αυτόν τον αγώνα και άρα να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινά φορολογικά έσοδα χάρη στη χρήση ορισμένων μέτρων που να καταλήγουν σε δικαιότερο ανταγωνισμό. Αλλά κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό έχει παγώσει φαίνεται και πρέπει η Κομισιόν να κάνει κάτι γι' αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω εδώ που λέμε τόσα μεγάλα λόγια ότι θέλουμε και Ευρώπη των έργων. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό κύριος Λάγκεν. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση για, την για τα φορολογικά θέματα δεν είναι ρουτινέρικη διαδικασία. Τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε πάντα αιτήματα για τη διαφάνεια και δεν έγινε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε να υπνώτει και οι εξελίξεις των τελευταίων μήνα κατέδειξαν πόσο αναγκαία είναι όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό χαιρετίζω αυτά τα πρώτα βήματα ιδιαίτερα, διότι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή έφτασε πια σε έναν όγκο που πραγματικά πλήττει τους έντιμους ε, φορολογούμενους εκατοντάδες εκατομμύρια ε, εργαζόμενους ε, και 20 εκατομμύρια τουλάχιστον μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν βλέπουμε ότι έχουμε ένα δις ετήσια, τότε κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη ήταν εκείνα τα οποία δεν οδηγήθηκαν σε αρμονισμό φορολογικό. Δεν πρόκειται για φορολογικό εναρμονισμό σε υψηλό επίπεδο, αλλά για μια στρατηγική αποκλειστικά κατά του φορολογικού dumping. Και σύμφωνα με το άρθρο 101 έως 109 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αθέμητος ανταγωνισμός και για φορολογικά θέματα απαγορεύεται. Σας ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κύριος Hayes. <clears throat> Θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε την επόμενη εβδομάδα είναι θετική. Καλωσορίζω το γεγονός ότι περνάμε σε βήματα προόδου στον τομέα της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών. Φυσικά και πρέπει να είμαστε κατά της επιθετικής φορολογικής πρακτικής, αλλά θα πρέπει βέβαια οι μεγάλες επιχειρήσεις να πληρώνουν αυτό το οποίο πρέπει. Δεν νομίζω όμως ότι απαιτείται και οι πολίτες επιθυμούν μια πλήρως εναρμονισμένη φορολογική πολιτική. <clears throat> Και αυτό φαίνεται στις εκλογές. Πρέπει να είμαστε αρκετά αυστηροί σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να φοροαποφύγουν συστηματικά. Εκεί πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Απαιτείται να γίνει και μία συζήτηση σε βάθος και εδώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, ουσιαστικά επίπεδα φορολογίας. Υπάρχουν ε, κάποιες χώρες που λένε ότι έχουν 30% αλλά το 30% στην ουσία δεν είναι αληθινό, είναι 8-9-10%. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι τα πραγματικά επίπεδα φορολόγησης και όχι τα τεχνητά. Ευχαριστώ. Κλείνει ο κατάλογος περνάω στο Catch the Μισή θα πάρουν το λόγο, έξι. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Καπούτο. ο κύριος Κέλλη μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Χέις. Εξέφρασε τη θέση μας γύρω από το θέμα αυτό, γύρω από αυτό τον φάκελο. Συμφωνούμε ότι η αποφυγή και η ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών είναι βασικά θέματα για να υπάρξει η δικαιοσύνη φορολογική και είμαστε υπέρ. Τις προτάσεις αυτές για το CCTV δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Ξέρουμε ότι σε ορισμένες χώρες υπάρχουν προβλήματα. Ε, νομίζω ότι ο ανταγωνισμός είναι κάτι το οποίο είναι υγιές γενικά και γιατί να μην υπάρχει και στον τομέα της φορολογίας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση αυτή λοιπόν και θα την καταψηφίσουμε όπως ακριβώς το κάναμε και στο παρελθόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Φλασίκοβα. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η φορολογική πολιτική έχει αγνοηθεί εν πολύ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα έχει θεωρηθεί ότι ήταν κάτι το δευτερεύον. Και αυτό νομίζω ε, υπογραμμίστηκε και από τη συζήτηση που έγινε σήμερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε να καταστήσουμε ε, σοβαρή την πολιτική μας τη φορολογία για να αποτρέψουμε την φοροδιαφυγή και να αποτρέψουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις να αναζητούν τις χώρες οι οποίες έχουν τους πιο, ε, τους, τις πιο ευνοϊκές ε, ρυθμίσεις. Στη Σλοβακία σαν παράδειγμα έχουμε χαμηλά επίπεδα φορολόγησης και βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ανταγωνισμός γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες σαν παράδειγμα οι οποίες έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες για φορολογικούς λόγους. Η κυρία Τόμασιτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αναγνωρίζεται η ανάγκη να μην υπερβαρυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με φόρους. Ωστόσο όμως πιστεύω ότι δεν έχει γίνει αυτό επαρκές γνωστό στα κράτη-μέλη σε σχέση με πολιτικές ε, για να ακολουθηθεί αυτή η πορεία επιτέλους. Πρέπει να καταπολεμηθεί η απάτη και η φοροδιαφυγή σίγουρα. Αλλά αυτό δεν θα είναι χρήσιμο αν τα κράτη-μέλη με τις διοικητικές δαπάνες και επιβάρυνση ε, υποστηρίζουν την μαύρη οικονομία, την παραοικονομία. Γι' αυτό πρέπει να πω ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία ανέφερε η συγγήτρια. Είπε η συγγήτρια κατά εκείνων των χωρών που υιοθέτησαν κάποια συστήματα ανταγωνιστικού χαρακτήρα και δεν φταίνε διότι φταίνε τα άλλα κράτη τα οποία έχουν απαρχαιωμένα συστήματα που λειτουργούν εκεί. Ευχαριστώ και εγώ πρόεδρε. Χαιρετίζω το περιεχόμενο αυτής της ετήσιας έκθεσης για τη φορολογία. Διότι αυτό είναι αυτό το οποίο χρειαζόταν μετά το σκάνδαλο LuxLeaks. Χρειάζεται διαφάνεια για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Μεγαλύτερο εναρμονισμό και <clears throat> συμμετοχή ώστε οι φορολογούμενοι να έχουν κάποιες δυνατότητες που θα προσαρμόζουν στην ίδια την πραγματικότητα. Η φορολογία πρέπει να εξυπηρετεί την ε, νόμιμη οικονομία και να μην υπάρχει δυνατότητα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και μάλιστα με επιθετικό χαρακτήρα. Και πρέπει να βοηθά με την καινοτομία και όχι τις αυταπάτες. Όσοι κάνουν τέτοια πράγματα κατά τα άλλα <clears throat> πέρα από τις κυρώσεις θα πρέπει να παραμείνουν στο περιθώριο όσον αφορά δημόσιες επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Χρειαζόμαστε τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ώστε να προχωρήσουμε και μια κατεπίγουσα μεταρρύθμιση του ΦΠΑ που είναι πεπαλαιωμένη η κατάσταση. Και στο τέλος συγχαρητήρια πρέπει να πω για την οικουμενική προσέγγιση, διότι αυτοί οι φιλοευρωπαϊστές αυτό επιθυμούν και αυτό θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, Βίγκα παρακαλώ. Eh, Αυτή η συζήτηση είναι πραγματικά μια αυταπάτη. Υπάρχει μεγάλη υποκρισία. Ο κύριος Γιούγκερ, για παράδειγμα, συνέζησε επί δεκαετίες με πρακτικές φοροδιαφυγές, και έδωσε κίνητρα και γι' αυτό. Είναι η κατάσταση πολύ ανησυχητική όσον αφορά την φορολογική δικαιοσύνη. Αυτή η έκθεση δεν είναι παρά ένα ευχολόγιο που δεν δεσμεύει κανένα. Αναφέρει σκάνδαλα, αλλά υπάρχουν, ε, θα έλεγα, ανέξω έξοδες διατυπώσεις που δεν θίγουν το πραγματικό πρόβλημα. Το πρόβλημα ανάγεται στη δεκαετία του 80, 1980 με την ε, φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη πολιτική δημιουργώντας ε, αυτοκρατορίες ε, εις βάρος της οικονομίας. Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, η διαφυγή και η φοροδιαφυγή είναι όλα αυτά πτυχές της ίδιας νόσου, της ίδιας ασθένειας και βλέπουμε εδώ πραγματικά όλα παραμένουν τα ίδια χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής από το ΚΑΤΣΔΙ, η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Στα θεωρία επίσης, μετά από τα σκάνδαλα LuxLeaks, όπου ο πρόεδρος Juncker της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως υπουργό Οικονομικών του ιδίου του Λουξεμβούργου είχε εμπλακεί, ο ίδιος υπεσχέθη ότι τώρα επιτέλους η φοροδιαφυγή θα πάψει να υφίσταται στην Ευρώπη. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για ένα μητρό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Αλλά δεν επαρκεί. Πόρο απέχει από το να επαρκεί. Χρειάζονται τώρα χρήματα που πρέπει να επενδυθούν στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στην, στον εξυγχρονισμό των συστημάτων μα. Και γι' αυτό <clears throat> στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δράσουμε. Και στη δική μου χώρα, την Αυστρία, είμαστε υπέρ του να αρθούν τα απόρριτα, τα τραπεζικά απόρριτα και όχι όπως το προτείνει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για κάποιους φορείς αλλά και για ιδιώτες. Είναι κατανόητο γιατί οι ιδιώτες μπορούν να φοροδιαφεύγουν με αυτόν τον τρόπο με τραπεζικό απόρριτο και πρέπει να δράσουμε. Πρόκειται για φοροαπάτη, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή μεγάλων διαστάσεων. Αυτό πρέπει να σταματήσει επιτέλους προς όφελος των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα κλείνει η συζήτηση και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Μοσκοβίση για να συνοψίσει. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σύντομα, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους σας για τη συμβολή σας στη συζήτηση. Κρατώ από αυτήν ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση περί των στόχων. Όλοι μας θέλουμε μια πιο δίκαια και πιο αποτελεσματική φορολόγηση στην Ένωση ένα διαφανές και προβλέψιμο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις μας και για την ανταγωνιστικότητά τους διεθνώς και θέλουμε οι διοικήσει των χωρών μελών να μπορέσουν να ασκήσουν καλύτερα τις δικαιοδοσίες τους που σήμερα έχουν αποδυναμωθεί. Αυτό το μήνυμα θα δώσουμε και εμείς και στους συναδέλφους μας και στις χώρες μέλη, στο Συμβούλιο δηλαδή να μην υπάρχουν κανόνες που κάνουν τα πράγματα πιο πολύπλοκα. Τρία σύντομα σχόλια τηλεγραφικά. Πρώτον, άκουσα παρατηρήσεις και ήθελα να σας πω ότι αυτό που προτείνουμε είναι ουσιώδες. Δηλαδή για τη διαφάνεια η πρόοδη της δέσμης που προτείνω αρχίζουν μια καινούργια εποχή χωρίς υπερβολή. Ποτέ δεν είχαμε προτείνει κάτι τόσο φιλόδοξο που ξεπερνάει κατά πολύ τα εργαλεία που έχουμε από το 77. Και προσθέτω ότι είναι βέβαια μία πρώτη φάση και όχι κάτι κάθε αυτό, δεν είναι αυτός σκοπός. Θα προτείνουμε δηλαδή μέτρα και ανταγωνιστικότητας και νέες φάσεις διαφάνειας. Μαζί σας θα τις εξετάσουμε καθώς και την ιδέα του country by country report. Αυτά που κάνουμε δεν τα κάνουμε για μας. Ζούμε σε παγκοσμιοποίηση σε συνεργασία με τον ΟΣΑ, με τις προτάσεις του Z20 και θέλουμε συνεργασία και με άλλες οντότητες πέραν της Ένωσης, παραδείγματος χάρη συγκρίνω με την συμφωνία για την τραπεζική αλληλοπληροφόρηση που θα υπογραφεί μέχρι το καλοκαίρι και αυτό είναι επανάσταση και θα καταργήσει στην ουσία το τραπεζικό απόρριτο. Τρίτον, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι αποφασισμένος να αλλάξω τα πράγματα γιατί και η κοινή γνώμη δεν ανέχεται πια ορισμένες αδικίες και πρακτικές και θέλουμε να θέσουμε τα κράτη-μέλη ενώπιον των ευθυνών τους. Και χρειαζόμαστε και εσάς βέβαια για να συνεργαστείτε με την Κομισιόν χέρι με χέρι και γι' αυτό θα προσέξω ιδιαίτερα όλες σας τις προτάσεις και γι' αυτό οι εργασίες σας εδώ παίζουν ουσιώδη ρόλο τόσο για την συνειδητοποίηση της κατάστασης όσο και για την πρόταση λύσεων και με ανυπομονησία τις προτάσεις αυτές και τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, η συγγήτρια κυρία Καϊλή τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε όλοι το λόγο. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου θέσαμε προτεραιότητες και θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε. Υπάρχουν κάποιοι τομείς τους οποίους δεν καταλήξαμε από κοινού, περιβαλλοντικά θέματα, παράγοντες που γεννούν απασχόληση, όπως επίσης και προστασία αυτών οι οποίοι δίδουν τις πληροφορίες, χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε τα στοιχεία που απαιτούνται. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο Μοσκοβισή για τη συνεργασία του μαζί μας και ζητάμε επίσης και από το Συμβούλιο να μας ακούσει. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα έχει μια σαφέστατη θέση, μια συνεκτική θέση. Ζητούμε εμείς μια ανταπόκριση στα προβλήματα αυτά η οποία να είναι φιλική στην επιχειρηματικότητα ε, να είναι φιλική με το περιβάλλον, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Καηλή. Τέλειωσε